Καλημέρα κυρίες και κύριοι και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι 9.35. Ας αρχίσουμε λοιπόν την ε, συνεδρίασή μας. Υπαριθμόν 1. Έγκριση της ημερησίας διαδάξεως, Αν έχετε σχόλια. Όχι. Καλώς. 2. Ανακοινώσεις Προέδρου. Πρώτα θα δώσω την ευκαιρία στους διερμηνείς να πούν ε, την ανακοίνωση. Ένα μήνυμα από του διερμηνεί. Βρισκόμαστε στην 24η μέρα των κινητοποίησεων και ακόμη δεν έχουμε δει κάποια αντίδραση εκ μέρου τη διοίκηση. Αντίθετα, ο Γενικό Γραμματέα κληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση του στη σημερινή συνεδρίαση Πολλοί συνάδελφοι από άλλε καμπίνε έχουν επιταχθεί και είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν. Σε ένδειξη αλληλεγγύη, η ελληνική καμπίνα δεν θα προχωρήσει σε στάση εργασία όπω αρχικά προβλεπόταν, ωστόσο η διερμηνία θα διακοπεί ακριβώ την προγραμματισμένη ώρα λήξη τη συνεδρίαση. Then... Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Α προχωρήσουμε στο υπαριθμόν 3 σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Θα ψηφίσουμε την έκθεση πρωτοβουλίας για την κατάσταση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. 387 τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Ο δε κύριος Μπροκ έχει συμφωνήσει τελικώς επί 45 συμβιβαστικών τροπολογιών. Υπάρχει και γνωμοδότηση της ΙΝΤΑ, άρθρο 54, και θα ε, ενσωματωθεί στο τελικό κείμενο. Ο κύριος Μπροκ, σε συμφωνία με τον κύριο Λάγκε, προτείνει προφορική ε, τροπολογία για να ε, ενταχθεί η γνωμοδότηση στην εκθεσή του. Α δώσουμε τον λόγο στον πρώην Πρόεδρό μας, κύριο Μπροκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ δηλαδή τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία και στην βάση της συνεργασίας αυτής νομίζω μπορούμε να αναμένουμε ευρεία πλειοψηφία. Υπάρχουν βεβαίως ε, και σημεία που θα μπορούσε κανείς να τα διατυπώσει διαφορετικά. εξετάζοντα τι ε, συμβαστικέ τροπολογίε. Τέλο πάντων σε ορισμένα υπάρχει πρόσημα μείον. Δεν νομίζω ότι είναι και καμιά καταστροφή. Το βασικό μου πρόβλημα για την έκθεση αυτή είναι εν ώψη των πολλών τροπολογιών να είναι τελικώς ευανάγνωστη η ε, η έκθεση και να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Ε, θα παρακαλέσω τη γραμματεία να ξαναδεί μετά τα κείμενα και με συμφωνία βέβαια με τους ε, σκιώδεις συγητές να βάλουμε κάποιες διευκρινιστικές τροπολογίες για την Ολομέλεια ώστε τελικό το κείμενο να είναι εύληπτο, να, είναι, να ρέει ομαλά. Ευχαριστώ λοιπόν και για τη συνεργασία με τη Γραμματεία και με τους σκιώδεις εισηγητές και εισηγητές. Κύριε Πρόεδρε, αυτά. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπροκ, άλλος κανείς? Θα ήθελε άλλος κανείς να λάβει το λόγο? Όχι. Τότε μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσως στην πολύ μακροσκελή αυτή λίστα ψηφοφοριών και αρχίζουμε εδώ, έτσι δεν είναι. Άρα, Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2, συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα τροπολογία υπάρχουν 65 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ Α, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρο. 126 πρώτα. 126 του κυρίου Επιτιδίου, του φίλου μα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Α επαληθεύσουμε πρώτη φορά. 131. Του κύριου Μπιουτικόφερ. Μια στιγμή, λέει ο πρόεδρος. Eric, Eric, there is a machine not working. Um, I'm voting in Ψηφίζω υπέρ, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν έχω 39 συνάδελφοι είναι παρόντες. Τώρα έχει τελειώσει η ψηφοφορία. Ισοψηφία 19-19, μία αποχή. Α, είστε υπέρ. Και το χαλασμένο μηχάνημα. Άρα, πάλι ισοψηφία, 20 προς 20 και μία αποχή. Άρα, εκπίπτει. Άρα, ε, απορρίπτεται, συγγνώμη. Απορρίπτεται. Καλό, λοιπόν, καλώς λοιπόν που την επαληθεύσαμε. Συμβαστική 10, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά αποχές. Θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε και εδώ. 140 το κύριο Μπιτικόφερ αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται αυτή 24-16. 141 γκόμιος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16. Είναι όμως συμβιβαστική παρόλο που δεν είναι με γκρίζο χρώμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 199 και 200 που είναι ταυτόσιμες φώτιγκα βίστησεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε 222. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται λοιπόν 23 υπέρ 17 κατά. 223 φώτιγκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λείπει ένας. Τέλος. Απεριφθεί αυτή εδώ. 18-21. 225, 226 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 231 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 232 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Ας το επαληθεύσουμε αυτό το δεύτερο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος, απερίφθη. 234 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται, έτσι δεν είναι. Εγκρίνεται. 243 σε δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται σαφέστατα. Συμβασία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 253 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 255 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 256 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, επαλήθευση 256 τμήμα δεύτερο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται με σαφέστατη πλειοψηφία. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 262 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αυτή εκπίπτει όμω, διότι εγκρίναμε το πρώτο τμήμα της προηγούμενης. Όμω τι σημαίνει αυτό. Για τον Nord είναι αυτό που λέτε. No vote, λοιπόν. Οκ. Okay. Τώρα, συμβαστική 27. Υπέρ, κατά, αποχές,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 για αυτό το subheading, κύριε Πρόεδρε, το οποίο ζητεί να υπερασπιστεί το εμπόριο σε βάση κανόνων σε καιρούς trouble times, σε καιρούς ε, αναταραχής. Λοιπόν, μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Έρχομαι τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 Καστάλντο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Όχι λέει κάποιος από κάτω. Στην δική μου λίστα είναι όντως σε δύο τμήματα λέει ο πρόεδρος. Μόνο ο κύριος είναι και άλλοι. Είναι και άλλοι. μην ξεκινήσετε επανάσταση. 25. Καστάλτο. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο, δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Καστάλτο. Πάλι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας την επαληθεύσουμε αυτήν εδώ την ψηφοφορία. 26 Καστάλτο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πρόκειται για την αιτιολογική σκέψη Β. Πέρας. 22 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31, αντρική 1, υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση, επαλήθευση.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην υπαριθμόν 8 ε, υπέρ λοιπόν, κατά 7 ε, αποχές απορρίπτεται. Δεν είναι αναγκαίο να ψηφιστούν τα υπόλοιπα που αναφέρονται στην γνωμοδότηση της Επιτροπής ΙΝΤΑ και φτάσαμε ήδη στην τελική ψηφοφορία. Ωραία. Φτάνουμε λοιπόν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο της ε, ε, εκθέσεως όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 35 ψήφους υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε τον εισηγητή.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 So, dear colleagues, ladies and gentlemen, we better continue. Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε. Και περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Σε συνεργασία με την Υποτροπή για, την ανθρώπινη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της κοινότητας των Άνδεων, ενημέρωση για τη συνοδευτική ε, αντιπροσωπεία στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Κολομβία. Συνάδελφοι, να σας παρακαλέσω όσους από εσάς θέλετε να συνεχίσετε την, ε, τη τις σας για τα αποτελέσματα των μάτς του Μουντιάλ τα χθεσινά βραδινά να φύγετε. Οι Ιταλοί δυστυχώς δεν πέρασαν στον επόμενο γύρο, ούτε καν. Οπότε σας παρακαλώ πολύ, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να κοροϊδεύετε τους Γερμανούς. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, η αντιπροσωπή αυτή παρακολούθησε και τους δύο γύρους ε, των εκλογών 27 Μαΐου και 17 Ιουνίου και επειδή δεν υπήρχε ολοκληρωμένη επίσημη αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπα, αυτό δεν επρόκειτο για μια αποστολή επίσημη εκλογικών αντιπροσωπών ε, παρατηρητών ε, απλά μια συνοδευτική αντιπροσωπεία όπως είπα. Θέλω να υποδεχθώ και να καλωσορίσω την ε, κυρία Μπαραντίκα την ε, πρόεδρο της ε, ad hoc αντιπροσωπείας αυτής καθώς και τον πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον κύριο Παντσάρη, που δεν είναι όμως εδώ καθώς και τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της κοινότητας των Άνδεων τον κύριο Πασκουάλ που ούτε αυτός είναι εδώ, δεν πειράζει ε, να μας πει λοιπόν η κυρία Μπαραντίκα τι συνέβη σε αυτήν την ε, επίσκεψη. Πρωτού όμως δώσω το λόγο, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα αν η Επιτροπή ΑΦΕΤ είχε συμμετάσχει πιο ενεργά στην προετοιμασία αυτή τη αποστολή. Καταλαβαίνω ότι είναι μια ad hoc απόφαση που έλαβε η Προεδρία. Παρ' όλα αυτά, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα μου επιτρέψει να πω ότι έχει την εμπειρογνωμοσύνη και θα μπορούσε να είχε συμβάλει θετικά στην επίσκεψη αυτή. Εν πάση περιπτώσει, δίνουμε το λόγο στην κυρία Μπαραντίκα για να μα ενημερώσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθώς έχουν μείνει λίγοι βουλευτές, θα ζητούσα να με ακούσουν όσοι έχουν απομείνει. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη και συνοπτική. Θα τα πω σχηματικά. Πρόεδρος, συνάδελφοι. Η κυρία Μπιλμπάου ζήτησε να αποδώσετε την απαραίτητη προσοχή όσοι έχετε απομείνει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε πριν να ξεκινήσω με αυτή τη σύντομη παρουσίαση της ε, παρουσίας μας στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα ε, της ε, Αποστολής Παρατήρησης των Εκλογών για την καλή δουλειά, για όλη τη συμμετοχή και για τα καλά αποτελέσματα τα οποία πετύχαμε χάρη της παρουσίας τους από τις 23 ως 29 Μαΐου παρευρεθήκαμε για τον πρώτο γύρο των εκλογών ε, όπου συναγωνίστηκαν έξι ε, υποψήφοι ο Ιβάν Ντούκε και ο Γουστάβο ε, Πέτρο ήταν τα δύο φαβοροί. Αυτοί οι δύο ήταν που πέρασαν στη δεύτερο γύρο, όμως προς έκπληξη όλων γιατί σε καμία δημοσκόπηση δεν έλεγαν κανένα αποτέλεσμα στο Σέχιο Φαρχάντο που ουσιαστικά ήρθε στην τρίτη θέση με διαφορά 261.000 ψήφους, 60.000 ψήφους ε, από το δεύτερο. Κέρδισε πολλές ψήφους ε, στην Μπογκοτά και μάλιστα λεγόταν ότι αν είχε περάσει το δεύτερο γύρο θα ήταν ο πρόεδρος της Κολομβίας από τις 15 ως τι τις 18 Ιουνίου ήμασταν παρόντες για το δεύτερο γύρο. Ο Σέρχιο Φαχάντο ζήτησε ε, από τους πολίτες να ψηφίσουν λευκό, όμως ε, στο δεύτερο γύρο ήταν ο Ντούκε που πήρε το καλύτερο αποτέλεσμα με 53,8% και ο κύριος ε, Πέτρο με 42%. Η συμμετοχή ξεπέρασε το 53%. Οι εκλογές για το Κογκρέσο είχαν συμμετοχή μόνο 49%. Ήταν ειρηνικές εκλογές και οι πολίτες φαίνονται χαρούμενοι που μπορούσαν να ψηφίσουν σε ειρηνική κατάσταση η συμφωνία που υπεγράφει από τα πολιτικά κόμματα ε, ε, στο σύμφωνο για τη μη βία βοήθησε στο ειρηνικό κλίμα. Ήταν οι συζητήσεις ε, σε δημόσιους χώρους. Όμως η εκστρατεία ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτη σε σημείο που η Βαν Ντούκε απέρριψε να κάνει μια συζήτηση με τον αντιπαλό του στη δημόσια τηλεόραση. Η προεκλογική στρατεία ήταν αρκετά πολλωμένη μεταξύ των δύο και φυσικά ο κεντρικός άξονας ε, ήταν ε, το θέμα της τήρησης ημής της συμφωνίας ο Ντούκε ανακοίνωσε τη δυνατότητα να γίνουν κάποιες προσαρμογή στη συμφωνία και αναγνώρισε τη συνταγματικό του χαρακτήρα. Ε, στο δεύτερο γύρο ε, συνεχίστηκε αυτή η συζήτηση. Ήταν η ενδιαφέρουσα συνάντηση με την αποστολή παρατήρησης των εκλογών που μας είπε ότι το επίπεδο των ε, λαθών δεν έφτασε ούτε καν στο 0,3% στον πρώτο γύρο. Η πιθανή νοθεία που ισχυρίστηκε ο Πέτρος ε, στον πρώτο γύρο επιλύθηκε και απαντήθηκε με τα κατάλληλα επιχειρήματα ότι δεν έλαβε χώρα. Είναι απαραίτητο να προσεγγίσουμε και τις ε, διάφορες ε, μεταρρυθμίσεις ε, προκειμένου να δούμε ποιες ακριβώς είναι οι ευθύνες των διάφορων θεσμών στην εκλογική διαδικασία δεδομένου ότι οι δικαστές πάρα πολύ αργούν για να επιλύσουν τα διάφορα προβλήματα. Ε, είχαμε διάφορους ε, συνομιλητές όπως η διαφάνεια για την Κολομβία, ε, την παρουσία των δικοστών, την ομάδα της μνήμης από την Επιτροπή της Αλήθειας, ε, ή την Διευθύντρια των Εξαφανισμένων. Ε, όλοι αυτοί συμμετείχαν στη διαδικασία. Όλοι αυτοί γνωρίζοντας, αναγνωρίζοντας τη βοήθεια των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργανών στην ειρηνευτική διαδικασία μας ζήτησαν να συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε ε, στην εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας και μας έδειξαν, μας τόνισαν κάποιες ανησυχίες σε σχέση με τη στάση του κυρίου Ιβάν που κέρδισε τις εκλογές. Αυτή είναι η σύνοψη στους ε, δύο γύρους και τη συμμετοχή αυτής της αντιπροσωπείας ε, ad hoc από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Thank you, Ms. Bilbao. Ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Οι κύριοι Παντζέρη και Δεγκράντες Βασκουάλα αποσιάζουν. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω αν άλλοι συμμετέχονται στην αποστολή θέλουν το λόγο. Κύριε Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε πέρα από την ε, στάση κάποιου μέλους ε, της αποστολής ε, που ανήκει στις ιστορίες του μαγικού ρεαλισμού, τον Καβριέλ Γαρσία Μάρκες. Θέλω να πω ότι η παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κοινοβούλιο αποτιμήθηκε πολύ θετικά, πέρα από κάποιες ελλείψεις στο εκλογικό σύστημα. Εμείς θεωρούμε ότι η διαδικασία ήταν πολύ διαφανής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε κάθε ευκολία για να ολοκληρώσει την αποστολή του, κάθε διευκόλυνση. Σε σχέση με άλλε χώρες, η Κολομβία είναι μια χώρα που δίνει ένα παράδειγμα κανονικότητας ως προς την οργάνωση των εκλογών. Φυσικά δεν υπάρχουν τέλειες εκλογές ε, και όλα τα συστήματα μπορούν να βελτιωθούν. Όμως το πιο σημαντικό στην εκλογική αυτή διαδικασία είναι ότι για πρώτη φορά οι ΦΑΡΚ ε, δεν απειλούσαν την εκλογική διαδικασία που μπόρεσε να υλοποιηθεί μετά από πολλές ε, δεκαετίες χωρίς την παρουσία αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Και νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε ότι είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, περίπου στο 56%. Η χώρα της οποίας θα προεδρεύσει ο κύριος Ντούκε είναι μια χώρα που έχει εξελιχθεί πάρα πολύ προς πάσα κατεύθυνση. Ο πρόεδρος έχει μια σειρά μεγάλων προκλήσεων να αντιμετωπίσει την εθνική συμφιλίωση σε μια πολλωμένη χώρα και φυσικά είναι ο πιο νέος πρόεδρος που, έχει η Κολομβία και θα πρέπει να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Πρέπει να κλείσει το διάλογο με τον ε, ΕΛΕΝ τις ε, σχέσεις ε, με τη ΦΑΡΚ και με τους γείτονες με τη Βενεζουέλα και φυσικά πρέπει να αντιμετωπίσει και τη μεταναστευτική κρίση. Και η δική μας επιτροπή αλλά και η ομάδα που ασχολείται με τον εκλογικό συντονισμό ζητήσαμε στην ύπατη ε, εκπρόσωπο να ε, οριστεί μια αποστολή παρατηρήση των εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δυστυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο, όμως η αποστολή του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μπόρεσε να υλοποιήσει το καθήκον της. Η Κολομβία έχει μια σειρά σημαντικών προκλήσεων οικονομική κατάσταση. Η χώρα αυτή είναι φίλος και τέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό η ε, επιτυχία ε, του νέου Προέδρου μας τονίζει ε, τα προβλήματα που έχει η χώρα, κοινωνικά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα. Ε, βέβαια έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια η χώρα, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι το κόμμα του κυρίου Πέτρο, ε, υποψήφιος αριστεράς, πήρε 8 εκατομμύρια ψήφους και εγώ ε, θεωρώ ότι ε, επειδή απέτυχε αυτός ε, ο πρόεδρος, ε, βλέπουμε ότι ακολουθείται μια λαϊκιστική οδός. Ε, εμείς βέβαια θα συνεργαστούμε με τις αρχές της Κολομβίας που εκλέχθηκαν από τις κάλπες. Και ουσιαστικά αυτό είναι το ισοζύγιο από πολιτική σκοπιά, πέρα από το πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε την αποστολή παρατήρησης των εκλογών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Αλλά συμμετέχοντας θα ήθελα κάτι να πει. Κυρία Λαλόντ. Παρεξήγηση από πλευρά μου. Θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω και πάμε στο σημείο 5 Μία ενημέρωση για την αποστολή στην Αρμενία στις 18 ε, Ιουνίου. Θα είμαστε σύντομοι. Λοιπόν, ad hoc αντιπροσωπεία στην ε, Αρμενία, 18 Ιουνίου, λίγο παραπάνω από ένα χρόνο από την τελευταία μας επίσκεψη στη χώρα. Εννιά μέλη συμμετείχαν, επικεφαλής ήμουν εγώ ως πρόεδρος της ΑΦΕΤ, μαζί μας είχαμε τον συμπρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest, τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Αρμενία, τον εισηγητή της Επιτροπής μας, τον κύριο Τόκες, καθώς και, τον, και την κυρία Σόφκο, την κυρία Τζιλ, την κυρία Θεοχάρου, τον κύριο Ζάλα και τον κύριο Αουστρεβίτσιους. Η αποστελή μας είχε πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Είχαμε μόλις μία μέρα για επισκέψεις. Ε, συναντηθήκαμε με τον νέο Πρωθυπουργό της ε, Αρμενίας, τον Πασινιάν, τον ε, Υπουργό Εξωτερικών, τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, τον Άρα Μπάμπλογιαν, με βουλευτές από όλα τα κόμματα Καθώ και τον ομόλογό μου, τον επικεφαλή τον πρόεδρο τη ε, πρόεδρο Εξωτερικών Υπηρεθήσεων. Πριν από τι συναντήσει μα αυτέ, συναντηθήκαμε και με οργανώσει Κοινωνία των πολιτών και με τον πρέσβη τη Ευρωπαϊκή Ένωση τον κύριο Σβιτάλκη. Εκδόθηκε και ένα δελτίο τύπου, το οποίο επικεντρωνόταν στα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίσαμε και είδαμε σε αυτή την επισκοπή. Να σα πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, συνεχάριμεν όλα τα, ομολόγου μα για την πολιτική μετάβαση, η οποία έχει ε, πραγματοποιηθεί χωρίς ε, αναταραχές και στο πλαίσιο του συντάγματος. Υπάρχει πολύ μεγάλη προσδοκία από την πλευρά του λαού της Αρμενίας για τις μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα. Εμείς επιμείναμε στην ανάγκη να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ε, σε συμφωνία με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και είπαμε ότι σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει βεβαίως πάντοτε να συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών και η αντιπολίτευση. Και βεβαίω, όπω είπαμε, για, είπαμε για τι επόμενε εκλογέ, ότι εμεί είμαστε έτοιμοι βεβαίω να έρθουμε ω παρατηρητέ. Για τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Αρμενία, του ενημερώσαμε για την ψηφοφορία που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια για την ολοκληρωμένη και ενισχυμένη συμφωνία εταιρική σχέση. Και εδώ ε, τονίσαμε τη σημασία τη εφαρμογή αυτή τη συμφωνία για να προσελκυστούν επενδύσει, για να προωθεί το εμπόριο. Επίση. ε, υποστηρίξαμε την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την κατάργηση των θεωρήσεων σε περίπτωση βεβαίως και υπό τον όρο μάλλον ότι θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες συμφωνίες και αφού αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των παρατύπω διαμενόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αρμενίων, που είναι ένα πρόβλημα σε πολλά κράτη-μέλη. Θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω βεβαίω όλου όσου συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, καθώ και τον πρέσβη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Σβιτάλκη, γιατί ήταν πραγματικά πάρα, πάρα πολύ σημαντική η συμβολή του. Ήταν πολύ λίγο ο χρόνο που είχαμε όλοι μα στη διάθεσή μου. Αυτά από την πλευρά μου. Πόσοι τέσσερι συνάδελφοι. Ε, είναι εδώ μόλις που πρέπει οπωσδήποτε να επανεκλεγούν σε επόμενες ευρωεκλογές. Θέλετε να προσθέσετε κάτι παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε ήταν μια πολύ χρήσιμη ε, και καλά προετοιμασμένη επίσκεψη. Είδαμε στην πράξη επιτόπου ότι η μετάβαση αυτή ε, κινείται ε, στη σωστή κατεύθυνση, έγινε με τον σωστό τρόπο. Ε, θα αποστείλουμε και παρατηρητές στις επικείμενες εκλογές και ο τροποποιημένος εκλογικός νόμος τη χάνει τις ικανοποίησεις και τις συμφωνίες όλων των πολιτικών κομμάτων. Γι' αυτό και στενά θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Αρμενία. Κατά τη γνώμη μου εκλογές δεν πρέπει να γίνουν αν δεν υπάρχει συμφωνία από όλα τα, κράτη, από όλα τα κόμματα που συμμετέχουν ε, ότι πράγματι τηρούνται οι συμφωνημένες κανόνες. Και πράγματι ε, ε, ε επιβεβαιώνω και εγώ ότι οι επίσημες αρχές της Αρμενίας ε, προσκάλεσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποστείλει παρατηρητές στις ε, εκλογές. Νομίζω ότι αν ακολουθούν όλοι οι κανόνες μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια σταθερή και ασφαλή διακυβέρνηση της χώρας. Ευχαριστώ. Ε, όχι, δεν έχω κάτι να προσθέσω. τα είπατε όλα, κύριε Πρόεδρε. Νίνα Γκίλ, ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι ήταν πραγματικά απίστευτη αυτή η επίσκεψη ήταν ταχύτατη ε, δεδομένων των πολλών συναντήσεων που είχαμε και πραγματικά ήταν ε, εντυπωσιακό να πας το ένα βράδυ στην Αρμενία να κάνεις 10 συναντήσεις και το επόμενο βράδυ να έχεις επιστρέψει ήδη στη βάση σου. Νομίζω ότι στο, στο, στο, στο μέλλον ήταν, ε, είναι, είναι θετικό να γίνονται τέτοιες επισκέψεις. Ήταν πραγματικά πολύ ωφέλιμη, πολύ χρήσιμη και μας έδωσε την ευκαιρία να σχηματίσουμε μια πολύ καλή εικόνα για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Αρμενία. Αυτό που κρατώ εγώ είναι ότι πραγματικά πρέπει να επιμείνουμε και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Αρμενία και να υποστηρίξουμε τους Αρμενίους και να ε, εξασφαλίσουμε ότι η Κομισιόν θα παράσχει τα απαραίτητα κονδύλια αλλά και την τεχνική αρρωγή που είναι απαραίτητη στη χώρα. Ε, δεν ξέρω αν μπορούμε κάποια στιγμή στην ΑΦΕΤ να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό, αλλά δεν θα ήθελα να το ξεχάσουμε έως τις επόμενες εκλογές. Ε, το συντομότερο δυνατό θα έλεγα, γιατί ε, αν οι εκλογές γίνουν ε, σε ένα χρόνο περίπου, δεν θα ασχοληθεί και κανείς, γιατί την ίδια περίπου περίοδο θα έχουμε και τις ευρωεκλογέ. Και αν πράγματι υπάρξει αποστολή παρατηρητών, δεν θα συμμετέχουν και πολλοί ε, ευρωβουλευτέ, όπω καταλαβαίνετε. Εκτό από του Βρετανού, βέβαια, που δεν θα έχουν να κάνουν ε, προεκλογικό αγώνα. Να πω επίση ότι με την ομάδα μου ε, παρακολουθούμε στενά τα πράγματα και την επόμενη εβδομάδα έχουμε και συνάντηση με το αδελφό κόμμα μα ε, που θα ε, μας επισκεφτεί στο Στρασβούργο. Συνεχίζεται λοιπόν ο διάλογο και θα ήθελα από αυτό το βήμα ε, να, τον, καλέσω και όλες τις άλλες πολιτικές ομάδες να ε, ενισχύσουν και να προωθήσουν τις σχέσεις τους με τα αδελφά τους κόμματα στην Αρμενία για να υπάρχει ένας καλός διάλογος με τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ και, και για την αποστολή όπως είπα και αρχικά. Ευχαριστούμε Νίνα, πραγματικά ήταν εξαιρετική η αντιπροσωπή αυτή, αυτή η επίσκεψη. Ε, ήταν πολυκομματική και με ενημέρωσε ο ε, ομόλογος μου, ε, ο πρόεδρος της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης τη Αρμενίας ότι ήταν πολύ μεγάλη προβολή μας και στα μέσα ενημέρωσης. Ωραία, περνάμε τώρα στο σημείο 6. Α, κύριε Λαλόν, με συγχωρείτε. Πιστεύω ότι έχουμε ένα πρόβλημα με την κατανομή του λόγου. Εγώ δεν συμμετείχα στην αποστολή στην Αρμενία, όμως ε, γνωρίζω αρκετά καλά την υπόθεση από την πλευρά του Αζερβαϊτζάν, ε, γιατί έχω πάει στον Αργόνο Καραμπάχ και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της σταθερότητας της Αρμενίας ε, και θα πρέπει να πιάσουμε για τις συμφωνίες του ΜΙΣΚ για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε αυτή την παγωμένη σύραξη που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αρκετά ανησυχητικά όσα είδαμε στην Αρμενία τα τελευταία, το τελευταίο καιρό. Έτσι λοιπόν ε, νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια δόση σταθερότητα. Um, Ευχαριστώ. Θα κάνουμε μια συζήτηση στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα για το θέμα της Αρμενίας, την Τρίτη το βράδυ. Οι συνάδελφοι θα μπορούσαν να ζητήσουν και εκεί το λόγο, γιατί πέρα από αυτή τη συμφωνία συνεργασίας θα συζητήσουμε και τη γενική κατάσταση και εξέλιξη της Αρμενίας. Πάμε στο σημείο 6. Θα ενημερώσουμε την Επιτροπή για την αποστολή μας ε, στο ΑΣΕΑΝ, στην Ινδονησία και στην Ταϊλάνδη από τις 8 11 ε, Μαΐου οργανώστηκε ε, μαζί με την αποτροπή ΤΑΖΕ η ε, αποστολή αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες Ανατολική Ασία και την ΑΣΕΑΝ. Επισκεφθήκαμε την Ινδονησία και την Ιλάνδη από τις 8 στις 11 Μαΐου. Θέλουμε να προωθήσουμε στρατηγικές σχέσεις με την Ινδονησία και την ΑΣΕΑΝ και να συνεισφέρουμε στην ε, ε, σταδιακή επαναδέσμευση με τον παραδοσιακό μας σύμμαχο την Ταϊλάνδη κατόπιν των συμπερισμάτων του Συμβουλίου του προηγούμενου Δεκεμβρίου και εν ώψη των μελλοντικών εκλογών. Είχαμε πολλές συναντήσεις στην Ινδονησία και στο ε, Γενικό Επιτελείο του ΑΣΕΑΝ ε, με τον έκτο πρόεδρο της Ινδονησίας, τον κύριο Σουσίλο Μπάμπανκ, τον σημερινό αντιπρόεδρο της Ινδονησίας, Γιούσεφ Κάλα, τον γενικό γραμματέα ΣΕΑΝ, τον κύριο Ντάτο Λιμ Τζοκχόη, τον ε, Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Ινδονησίας, τον κύριο Μασούρτη και τον ε, αναπληρωτή πρόεδρο της Βουλής Φαρτισών. Στην Ταϊλάνδα συναντήσαμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Φρακτρούλε, τον ε, πρώην Πρωθυπουργό του Δημοκρατικού Κόμματος και τον ε, πρώην, ε, τους πρώην αντιπρόεδρους της κυβέρνησης ε, Τσάισαν και Τεπ Καντζάνα και τον πρόεδρο της Βουλής. Ενημερωθήκαμε για την κατάσταση διμερών σχέσεων, τα τρέχοντα θέματα που πρέπει να επιληθούν και την ε, μακροπρόθεσμη αξία αυτών των εταίρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπούμαστε ότι ε, τόσο πολύτιμες μελλοντικέ εταιρικέ ε, σχέσεις επισκιάζονται από άλλα θέματα όπως πολλαπλές κρίσεις στην άμεση γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συναντήσαμε πολλούς εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών από ε, από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, μέχρι και υπερασπιστές του περιβάλλοντος. Ε, επίσης είχαμε συναντήσεις με τα κύρια πολιτικά κόμματα στην Ταϊλάνδη θα ήθελα να αναφέρω, είχαμε κάποιες συναντήσεις κλειδιά στην Ινδονησία με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Αντιπρόεδρο που όμως επισκιάστηκαν από τις ανησυχίες της Ινδονησίας σε σχέση με το έλεο ε, στα μελλοντικά πρότυπα βιοκαυσίμων ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Ινδονησία επίση συζητήσαμε την κρίση του προσφυγικού στην Μιανμάρ και αποφύσαμε να περιλαμβάνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ατζέντα του ΑΣΕΑΝ. Στην ε, Ταϊλάνδη θα ήταν καλό να μπούμε σε ένα ανοιχτό διάλογο παρά να απομονώσουμε αυτό το σύμμαχο στην Τελική Ασία. Ε, υπενθυμίσαμε στις αρχές Ταϊλάνδης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εμβαθύνει τις διμερείς σχέσεις ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπογραφεί η Συμφωνία Εταιρική Σχέση και να διαπραγματευτούμε μια Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, ε, αλλά όλα αυτά υπό ελεύθερες και δίκαιες και αξιόπιστες εκλογές οι εκλογέ προβλέπονται για το Φεβρουάριο του 19, αλλά ίσω να καθυστερήσουν ε, αν δεν έχουν περάσει τα απαραίτητα εκλογικά νομοσχέδια ε, ή αν αποφασίσει αλλιώς ο στρατός. Όμως υπάρχει η αν αποφασισει αλλιώ ο στρατό. Όμω υπαρχει η λαικη πιεση να γίνουν οι εκλογές ε, το συντομότερο. Κατά τη διάρκεια τη συνάντησή μας ε, με την Εθνοσυνέλευση, με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευση, εκφράσαμε την επιθυμία μας να δούμε μία παρατήρηση, αποστολή παρατήρηση των εκλογών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο στις εκλογές του χρόνου. Υπενθυμίσαμε ότι θα πάμε μόνο μας προσκαλέσουν και αν οι εκλογές είναι αξιόπιστες και υπάρχει ε, μια θετική δήλωση από την αποστολή παρατήρησης των εκλογών αυτό θα ωφελούσε την Ταϊλάνδη και τη φήμη της ε, στην προσπάθειά της να ε, επανα συστήσει τι στενέ διεθνεί σχέσει. Η αποτελεί μα από την ΑΦΕΤ αποτελούνται από του ακόλουθου συναδέλφου Πρέντα, Ζόφκο, Φρουντζουλίκα, Λόπε Αγγιλάρ, Καν, και ΠΑΕΤ. Και είχαμε συναδέλφους από την ΑΣΕΑΝ. Αυτά από μένα. Σχόλια από τη δική σας πλευρά. Σοφκόχη, Μπούχνα. Δεν βλέπω άλλο παρόντα. Επομένως πάμε στο επόμενο θέμα, διάφορα. Δεν υπάρχει νομίζω κάτι. Η επόμενη συνεδρίαση 9 Ιουλίου από τις 3 στις 6.30 το απόγευμα και 10 Ιουλίου από τις 9 στις 12.30 και 2.30 μέχρι 6.30 το απόγευμα. Ολοκληρώνει τη συνεδρίασή μας.